κόσμο. Ο ανταγωνισμός για τη γνώση σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι. Έληξε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, την Τετάρτη, ε, συγγνώμη, μεθαύριο Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Μορέρα με θέμα εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή δεν εκπονήθηκε από μένα προσωπικώς μόνον. Είμαι ένα πληρωτής εισηγητής, διότι ο αρχικός εισηγητής εγκατέλειψε την έκθεση και εγώ ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, της Αρμόδιας, ακολουθώντας τους κανόνες, ανέλαβα την ε, έκθεση. Είμαι και ένας ε, υποχρεωτικός εισηγητής γιατί δεν υπερψήφισα την έκθεση και έχω και σοβαρές ενστάσεις. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα και δυστυχώς ε, αναλαμβάνω ε, την έκθεση αυτή. Όπως γνωρίζουμε αυτή η έκθεση για την εκχώρηση ειδικών ε, εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν προέκυψε από απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια πρόταση. Επειδή ακριβώς ε, πρόκειται για έκτακτης ανάγκης εμπορικές προτιμήσεις, οι οποίες ε, δεν συνάδουν με τον κανόνα της θετικής ή αρνητικής ε, διάκρισης του ΠΟΕ, θα πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει μια απαλλαγή από τον ΠΟΕ, ώστε αυτές οι εμπορικές προτιμήσεις να γίνουν αποδεκτές. Έγινε βέβαια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και ε, η Επιτροπή Ίντε, της οποίας είμαι πρόεδρος, ε, εξέτασε την έκθεση και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με συζήτηση και ψηφοφορία. Και σας παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το θέμα, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν ε, αντικείμενο διχογνωμίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Τόσο Όσον αφορά το γεγονός ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, εμπορικές προτιμήσεις ως ε, μέσο κατεπίγουσας βοήθειας σε μια συγκεκριμένη χώρα και αυτός ήταν και ο λόγος ε, για τον οποίο έγινε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τη διάρκεια αυτών των εμπορικών προτιμήσεων και την επέκτασή τους και συζητήθηκε επίσης και το θέμα των όρων που θα πρέπει να τεθούν από τη χώρα που θα επιφεληθεί από αυτές τις προτιμήσεις, το Πακιστάν εν προκειμένου. Υπερψηφίστηκε μεν ε, η δυνατότητα αυτών των εμπορικών προτιμήσεων ε, για το Πακιστάν. Στην πραγματικότητα όμως η Επιτροπή ε, ψήφισε και αρκετές τροπολογίες οι οποίες θέλουν να περιορίσουν τις συνέπειες αυτών των εμπορικών προτιμήσεων που θα εκχωρηθούν στο Πακιστάν. Και μεταξύ των τροπολογιών υπάρχει και μία ρήτρα διαφύλαξης εάν ε, ε, υπάρξει μεγάλη απότομη αύξηση των ε, προτιμήσεων για το Πακιστάν και υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες αφορούν το γεγονός ότι το Πακιστάν δεν ήθελε να άρει τους περιορισμούς που επιβάλλει για τις εισαγωγές. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η προσπάθειά μας θα μπορούσε να αποβεί άκαρπη εάν δεν γίνει αποδεκτή από τον ΠΟΕ καταρχάς και ε, ε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα υπάρξει αποδοχή. Παρά το γεγονός αυτό όμως, ε, πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία να κατανοήσουμε λίγο την έννοια και τα όρια της χρήσης ενός μέσου όπως αυτού, αυτό για να δώσουμε μια έκτακτη βοήθεια ή και μια κάποια πολιτική αποζημίωση σε μια χώρα όπως προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να δημιουργηθούν επικίνδυνα προηγούμενα σε αυτή την περίπτωση και να γίνουν πολιτικό μέσο οι εμπορικές προτιμήσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να είναι πιο αντικειμενικές και συγκυριακές ε, σε σχέση με τη χρήση τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Μορέρα, ε, τώρα το λόγο θα πάρει η Επίτροπος η κυρία Κρός, η οποία αντικαθιστά τον αρμόδιο Επίτροπο τον κύριο Ντεγκούχτ. Θα μας συναντήσει ο κύριος Ντεγκούχτ στο κλείσιμο της συζήτησης. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο εσείς. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε σήμερα νομοθετική πρόταση κατεπηγουσών προτιμήσεων για το Πακιστάν. Πρόταση που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ε, σαφή αίτηση του ε, Συμβουλίου των Υπουργών μετά από τις περσινές πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν και που προκάλεσαν ευρύτατες καταστροφές στην χώρα αυτή και στον κατοίκους της. Ευχαριστώ τον εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, Διεθνούς Εμπορίου, για, το, για την έκθεση. Προτείνει η Επιτροπή για 75 εξαγώγημα προϊόντα από το Πακιστάν προσωρινή μείωση ή κατάργηση των δασμών που θα απελευθερώσουν δηλαδή συνολικά περίπου το 1 τέταρτο των εξαγωγών του Πακιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για δύο χρόνια με μια ενδεχόμενη παράταση κατά ένα έτος ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι τέτοιου είδους εμπορικές παραχωρήσεις και ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως τα υφαντουργικά προϊόντα ενδέχεται να έχουν επιπτώσει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Γι' αυτό διασφαλίσαμε την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της κάλυψης των αναγκών του Πακιστάν και της διαφύλαξης των συμφερόντων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός προϊόντων που έχουν επιλεγεί είναι περιορισμένος. Βάλαμε όρο φύ στην απελευθέρωση των προϊόντων αυτών. Η απελευθέρωση αυτή θα είναι επίσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Στο μεταξύ ζητήσαμε επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να μας παραχωρήσει άρση της ισχύω των κανόνων του ΠΟΕ ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προτινόμενα μέτρα. Και όπως γνωρίζετε εξακολουθούμε να συζητούμε το θέμα αυτό και με άλλα μέλη, άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ και ελπίζουμε να καταλήξουμε σύντομα σε κάποια λύση. Οι εικόνες που είδαμε ανθρώπων που έχουν χάσει πάνη είδος βιοπορισμού έχουν ε, βεβαίως εγγραφεί στο μυαλό όλων. Δεν θα πρέπει ωστόσο να λησμονούμε και το τεράστιο κόστος εκείνων των καταστροφικών πλημμυρών και σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που ε, χρειάστηκε να δοθεί, αλλά και σε ό,τι αφορά την καταστροφή που προκάλεσαν. Αυτά τα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι από μόνα τους και έρχονται επιπρόσθετα από την σημαντική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια της τάξης των 180 εκατομμυρίων ευρώ που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πακιστάν. Παρά τα αυτά, φιλόδοξα εμπορικά μέτρα είναι και ουσιώδους σημασίας για να υπάρξει ουσιώδης ανάπτυξη της οικονομίας του Πακιστάν και θα πρέπει να είναι και τμήμα της μεσοπρόθεσμης ανταπόκρισής μας σε αυτές τις χωρίς προηγούμενο καταστροφές. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τις προτάσεις μας. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν προταθεί από μέρους σας. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες όλων αυτών των ε, τροπολογιών, οι πιο σημαντικές είναι οι Γνωρίζω ότι υπάρχει επιθυμία να επιβληθούν όροι σε ό,τι αφορά τον σεβασμό πλευρά του Πακιστάν ορισμένων θεμελιωδών αρχών. Κατανοώ τι ανησυχίε των προσώπων που έχουν καταθέσει τι τροπολογίε αυτέ και βεβαίω τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρο των σχέσεών μα από μακρού χρόνου με το Πακιστάν. Ωστόσο, λόγω του επίγοντου προσωρινούμενου χαρακτήρα των μέτρων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοιου είδους επιβολή όρων δεν θα ήταν σωστή. Ο διάλογος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της ε, συμφωνίας συνεργασίας μας με το Πακιστάν είναι εκείνη το πραγματικό πλαίσιο που πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά για να μπορέσει να καταλήξει η προσπάθεια αυτή και σε λύσεις με διαρκή μόνιμο χαρακτήρα. ώστε και να μην επιβάλλονται δασμοί ή άλλα ανάλογα αποτελέσματος μέτρα στις εξαγωγές, διότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε σοβαρά την εκχώρηση των προτιμήσεων, υποσκάπτοντας έτσι και το νόημα, το πνεύμα δηλαδή και το γράμμα του κανονισμού μας. Το ΔΕ Πακιστάν πρέπει να λάβει μέτρα που να είναι ευθέως ανάλογα με τις διεθνείς υποχρώσεις του. Ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την επιβολή ορίων σε αφορολόγητα είδη από το Πακιστάν δεν θα πρέπει να ξεπερνά ορισμένα επίπεδα. Συμφωνώ επίσης ότι οι προτιμήσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν για οποιοδήποτε προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις ε, σε κάποιον Ευρωπαίο παραγωγό, εφόσον πρόκειται για παρόμοια προϊόντα και αυτό μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επίσης με ένα μηχανισμό επιβολής τελωνιακής εποπτείας και αυτό με τρίμηνες εκθέσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα σήμαινε υπερβολική ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση για τη χορήγηση αδειών κλπ και σε ό,τι αφορά την χρονική διάρκεια των εμπορικών προτιμήσεων θα είναι ε, ένα χρόνο από τη στιγμή που λαμβάνει ε, ε, μπαίνει σε ισχύ. Αυτό όμως νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει, είχε προτείνει μάλλον να ληφθούν τα εξαιρετικά αυτά μέτρα για μια τριετία. Το Συμβούλιο την περιόρισε σε δύο έτη με δυνατότητα παρατάσεως κατά ένατος ακόμη. Ωστόσο, να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διάρκεια των προσωρινών μέτρων σε ένα μόνο έτος θα σημαίνει ότι τα μέτρα πλέον στερούνται νόηματος. Σημειώνω επίσης ότι ο συμβασμός της 10 η Νοεμβρίου στο Συμβούλιο ήταν και για υφαντουργικά προϊόντα συμβασμός που εξαρτάται και από την εκ των υστέρων χωρίς έγκριση του ΠΟΕ για την άρση των δασμών αυτών. Μετά από την διαβούλευση αυτή, τα μέλη του ΠΟΕ ενδέχεται να επιβάλλουν και άλλα προϊόντα σε τέτοιες επιβαρύνσεις. Θα χρειαστεί λοιπόν να δούμε την άρση που θα χορηγήσει ο ΠΟΕ όταν θα έρθει αυτή. Σας διαβεβαιώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει αναέτος μελέτη επιπτώσεων για τις αυτόνομες προτιμήσεις που χορηγούνται στο Πακιστάν και θα υποβάλει τη σχετική έκθεση και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ακόμη λόγο για να υποστηρίξετε το μέτρο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνεργασία του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εγκριθεί η πρόταση αυτή μέσα σε ένα πνεύμα υπεύθυνη συνεργασία απέναντι σε χώρε που βρίσκονται σε ανάγκη. Κύριο για δύο λεπτά. E uh, Κυρία Πρόεδρε, μου φαίνεται ότι είναι πολύ σωστή η στιγμή κατά την οποία συζητούμε την έκθεση Πρέντα. Διότι Τώρα, αυτή τη στιγμή ακριβώς, συζητούμε τις εξαιρέσεις που ζητάει η Ένωση από τον ΠΟΕ. Είναι λοιπόν σημαντικό να δηλώσουμε, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους εμπορικούς μας εταίρους. Πρέπει η Ένωση να επιδείξει ότι είναι αποφασισμένη να χορηγήσει πρόσθετη και πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια από είναι είχε αποφασιστεί προηγουμένως για να επιτραέψει για να επιτραπεί η ανάπτυξη της πακιστανικής βιομηχανίας. Φυσικά για αυτά χρειάζεται χρόνος και πρέπει οι εμπορικοί εταίροι μας να το αναγνωρίσουν και αυτοί. Προς στιγμήν τα αποτελέσματα είναι αβέβαια, αλλά όπως δείχνουν και οι πρόσφατες εξελίξεις, είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε ένα σταθερό και ευημερών Πακιστάν χωρίς εξτρεμισμούς για να μπορέσει να αποδειχθεί αξιόπιστος εταίρος και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που δέχτηκαν τα περισσότερα από τα επιχειρήματα της Επιτροπής μας στη γνωμοδότησή της. Υπάρχουν όμως ακόμη δύο στοιχεία που για μας την Επιτροπή επέξουν ιδιαίτερα σημαντικά. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη σύνδεση μεταξύ των εμπορικών αυτών σχέσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων και των κοινωνικών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό θέμα και σημαντικό τμήμα όλων των συμφωνιών μας με το Πακιστάν και επομένως ακόμα και οι εμπορικές προτιμήσεις πρέπει να προϋποθέτουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Πακιστάν. Από την άλλη δεν έχει γίνει πλήρης αποτίμηση από την Κομισιόν των μέτρων αυτών και πρέπει άρα να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους στη ζωή του πληθυσμού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση στο Πακιστάν ακόμη και σήμερα μετά από εννέα μήνες εξακολουθεί να είναι άσχημη μετά από εκείνες τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Σωστά λοιπόν έδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και διέθεσε σημαντικά πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας πολλών εκατομμυρίων. Προσωπικά από την αρχή δεν ήμουν ικανοποιημένο για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από πίεση του Συμβουλίου πρότεινε και χρήση μηχανισμών του εξωτερικού εμπορίου για να δοθεί ενίσχυση στο Πακιστάν. Εγώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή αυτό το είπα κατ' επανάληψη και παρακάλεσα επίση κατ' στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή όσοι είναι αρμόδιοι για την άσκηση εξωτερική πολιτική και ιδίω η ύπατη εκπρόσωπο να έρθει στην Επιτροπή μα για εν πάση περιπτώσει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξηγήσει για ποιο λόγο θα πρέπει η βοήθεια αυτή να δοθεί μέσω του εξωτερικού εμπορίου. Να υπάρξει δηλαδή μια συνολική στρατηγική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή να μα εξηγηθεί, να ενταχθεί σε ένα κοινό πλαίσιο και να κάνουν προσπάθεια να μα πείσουν ότι αυτό έχει πραγματικό νόημα. Εξωτερικό εμπόριο για να δώσει μια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι Νταβίτ και, και άλλοι μπόρεσαν να φτιάξουν μια δέσμη η οποία βρήκε σημαντική πλειοψηφία μέσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Χαίρομαι επίσης για τον χρονικό περιορισμό των μέτρων, διότι μόνο έτσι μπορούν να αποφευθούν ενδεχόμενα σφάλματα. Όμως, ποια είναι η κατάσταση στο Πακιστάν τώρα. Έχει εξοδετερωθεί μεν ο Μπιν Λάντεν, αλλά το ερώτημα εξακολουθεί να εκκρεμεί, εάν δηλαδή και μέλη της κυβερνήσεως του Πακιστάν γνώριζαν περί της παραμονής του εκεί. Πολλοί από την ομάδα μου δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την ε, κατάσταση αυτή. Και δεν ξέρουμε επίση εάν οι άλλε χώρε μέλη του ΠΟΕ θα συμφωνήσουν και θα δώσουν την έγκρισή του. Καλό θα, θα ήταν λοιπόν αύριο να ψηφίσουμε τι τροπολογίε, ωστόσο να μην ψηφίσουμε σε τελική ψηφοφορία το ίδιο το κείμενο του ψηφίσματος, αλλά να το αναπέμψουμε εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε εάν χρειάζεται να μελετηθεί ακόμη. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ε, κύριε, κύριε Επίτροπε, Πραγματικά δεν κατανοούμε γιατί η πλειοψηφία της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου θέλησε να συζητήσει αυτό το θέμα για να ζητήσει αναβολή στη συνέχεια, κάτι με το οποίο διαφωνούσαμε. Είναι λανθασμένες και οι δύο αποφάσεις, αλλά και για χρονικούς περιορισμούς ε, θέλω να σταθώ μόνο στην ουσία να σας πω όμως ότι συμφωνώ απολύτως με την παρέμβαση του Προέδρου Βιτάλ Μορέια. Σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ε, καθημερινά πλήττεται από πολλές τραγωδίες, ε, φυσικές και μη, θα δημιουργήσουμε πολύ σημαντικό προηγούμενο εάν κάθε ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη γίνει ε, δυνατότητα εμπορικών προτιμήσεων. Θα δημιουργηθούν ανισότητες ε, προς ε, φτωχότερες χώρες και μόνο μέσω ισορροπημένων και διαρκών κανόνων μπορεί να υπάρχει όφελος για αυτές τις χώρες ε, που δεν μπορεί να υποκαταστήσουν τις εμπορικές προτιμήσεις με τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Δεν θα υπάρχουν πλέον εκτήματα για τους πλημμυροπαθείς που χτυπήθηκαν ήδη εδώ και ένα χρόνο στο Πακιστάν μόνο ο τομέας της ευρωπαϊκής κλωστοϊφαντουργίας θα πληρώσει το τίμημα αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής και ε, δεν θα πρέπει να έχουμε παρεκκλήσεις ε, στους εμπορικούς κανόνες χωρίς να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες ε, στα επιχειρήματά μας. Εάν θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη στους πληθυσμούς που πλήχθηκαν από τις πλημμύρες θα έπρεπε να αποφασίσουμε να βοηθήσουμε ώστε και να μην ε, ε, υποβοηθήσουμε την δέσμευση του Πακιστάν και τα όσα βλέπουμε σήμερα ε, για τον Μπιν Λάντεν δείχνουν ότι δεν είναι αξιόπιστη η χώρα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και τα θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία προέκυψαν προσφάτως. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Ρινάλντι για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι δεν πάει καλά σε μια συζήτηση που γίνεται το Μάιο του 2011 και αναφέρεται σε μια φυσική καταστροφή του καλοκαιριού του 2010. Μια φυσική καταστροφή που άφησε 12.000 ανθρώπους χωρίς ε, κατοικία και κατέστρεψε, συγγνώμη, 12 εκατομμύρια και ε, κατέστρεψε τις κατοικίες τους. Αυτή τη στιγμή διστάζουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνδράμουμε το Πακιστάν και το γεγονός ότι δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα ε, μας προσθέτει και το γεγονός ότι ε, δεν έχουμε πιο όρημη ε, εικόνα για την εμπορική πολιτική. Η εμπορική πολιτική θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των μέσων για να βοηθήσουμε λαούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι έχει δράσει καλώς ε, και σύντομα ε, και υπάρχει ένα πακέτο το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε για να μην τιμωρήσουμε ε, κάποιους τομείς οι οποίοι ήδη πλήττονται από την κρίση. Εμείς υποστηρίζουμε την τροπολογία 37 που επιτρέπει και στις επιχειρήσεις να ζητήσουν εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης είναι χαλεπή η καιρή αυτή για το Πακιστάν και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ζητούμε από την Ινδία να αλλάξει στάση και να ε, μην αρνείται συστηματικά τα ε, την, ε, την ε, άρνηση βοήθειας στον ΠΟΕ. Φυσικά υπάρχουν δυσκολίες στη σχέση μεταξύ των χωρών αυτών. Υπάρχει και η απόπειρα στη Βομβάη και το γεγονός ότι δεν συμμετείχε το Πακιστάν στη σύλληψη των δραστών αυτής της απόπειρας. Αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει και στοιχείο ρήξης επειδή ακριβώς υπάρχουν κακές σχέσεις γειτονίας. Ζητάμε βέβαια και από τις αρχές του Πακιστάν να είναι πιο αποφασιστικοί και να εφαρμόζουν και διμερώς κάποια θέματα θέματα και να συζητηθεί το θέμα διμερώς με την Ινδία. Έγιναν διμερώς οι συζητήσεις και δυστυχώς λίγα προέκυψαν από τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι το Πακιστάν και η διπλωματία του κρίκετ ε, την οποία μας επισήμαναν οι συνάδελφοι από το Πακιστάν με τους οποίους ε, συναντηθήκαμε πριν από κάποιες εβδομάδες δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως κάναμε και στη Γενέβη στην πρόσφατη διακευβουλευτική συνέλευση, ζητήσαμε να εφαρμοστούν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα επιτρέψουν στο διεθνές εμπόριο να ανταποκριθεί ταχύτατα στις κατεπίγουσες ανάγκες μιας χώρας η οποία πλήχθηκε από αυτή την καταστροφή. Το θέμα αυτό με τον δασμό θα μπορούσε ίσως να αποβεί ένα μεγάλο μηδενικό ή να δημιουργήσει μια νέα εποχή για τις εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Mr. President, Commissioner, colleagues. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Πρόκειται για τη χειρότερη θεομηνία που έπληξε ποτέ το Πακιστάν. Με περηφάνεια μπορούμε να πούμε ότι αντιδράσαμε γρήγορα. Η Επίτροπος Γεωργίευα πήγε επί τόπου και όταν συνάντησα και εγώ τον Πρωθυπουργό Ιουσούφ Ρεζαγκυλάνη μπορέσαμε να δούμε μου είπε και εκείνο πόσο επαρκής ήταν η ανταπόκριση της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πέρα από προκαθορισμένες γραμμές να βρούμε λύσεις όχι μόνο σαν την χορήγηση βοηθείας αλλά και εμπορικά μέτρα. Χαίρομαι γιατί η Επιτροπή δέχτηκε μετά από πολλές συζητήσεις και μετά από τη σκληρή δουλειά πολλών συναδέλφων ένα κείμενο κοινά αποδεκτό. Φοβάμαι όμως ότι μερικές από τις τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε ήδη ο Επίτροπος έχουν καταστρέψει ή μειώσει, αλλοιώσει το πνεύμα με το οποίο αρχικά θέλαμε να αντιδράσουμε. Έχουν ακουστεί αντιρρήσεις ήδη για τις προτάσεις μας που έλεγαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ της δράσης της Ένωσης και της ΕΖΕ σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει μία αντίφαση αν λέμε κάτι τέτοιο και ταυτόχρονα μιλάμε για άμεση σχέση με το Πακιστάν. Ταυτόχρονα όμως έχουμε την εγγύηση των αιτήσιων αξιολογήσεων. Καταλαβαίνω τι εννοείται για τα προβλήματα ασφαλείας, αλλά και εγώ είμαι από εκείνους που μόλις και επέζησαν τις επιθέσεις της Βομβάης. Και γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τώρα ώρα να ξεχάσουμε το Πακιστάν. Υποστηρίξτε τις προτάσεις. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Όλοι ξεπεράσατε το χρόνο σας. Πολύ. Σας παρακαλώ λοιπόν να τον σέβεστε στο εξής. Των πρασίνων για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ και άλλοι συμφωνούμε ότι τα θύματα των τρομερών πλημμυρών στο Πακιστάν είναι κάτι με το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, ως προς το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε όλοι μας την ελληνική. Αλλά ο ΠΟΕ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να χορηγήσει βοήθεια. Υπάρχουν όντως τροπολογίες που όντως αλλοιώνουν το πνεύμα της πρότασής μας και επειδή είναι επίγον να χορηγηθεί η εξαίρεση και να μειωθεί από τα τρία χρόνια στο ένα, στο ένα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο Πακιστάν να υφίσταται χαμηλότερους δασμούς. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τις συστάσεις αυτές είναι κάτι που δημιουργεί απλώς πρόσθετη γραφειοκρατία. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Συμφωνώ, καταλαβαίνω, κατανοώ το πνεύμα των προτάσεων που ζητούν αναπομπή στην Επιτροπή, η τροπολογία 43 δηλαδή, αλλά πότε θα έχουμε μια πρόταση που πραγματικά να μπορεί να επιφέρει πραγματικά αποτελέσματα στην πραγματικότητα που ζει το Πακιστάν. Πρέπει να δούμε πώς εργάζεται ο ΠΟΕ και να κάνουμε προτάσεις για να μετατραπεί σε πραγματικά δημοκρατικό οργανισμό με διαφάνεια και με μέλη που να λογοδοτούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και περίπου ένα χρόνο πλήγει το Πακιστάν από καταστροφικές θεομηνίες. Το σκάνδαλο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ ακολουθούν και αυτό δείχνει ότι αυτές οι εμπορικές διευκολύνσεις δεν είναι κατάλληλο μέσον για τη χορήγηση ενίσχυσης. Η πολιτική μου ομάδα έχει ζητήσει κατ' επανάληψη να υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο ώστε να ενισχυθεί ο λαός του Πακιστάν για την ανοικοδόμηση της χώρας του. Ποτέ ωστόσο δεν υποβλήθηκε μια εναλλακτική πρόταση. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στερείται ιδεών διότι οι αντιστάσεις του ε, Συμβουλίου τις είναι γνωστές. Φαίνεται πάντως οι δύσκολες διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να χρησιμοποιούνται ως άλοθη για την αδράνεια της Κομισιόν. Όμως αυτά τα ήξερε και από πριν. Ήδη δηλαδή όταν ορισμένοι υπουργοί και της Ομοσπονδιακής Γερμανίας έστειλαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα κάνει, να ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τα, ε, να προτείνει τα μέτρα αυτά. Ενώ άλλα Άλλες χώρες όπως η Μπαγκλαντές επέτυχαν σημαντικές συμφωνίες και μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Το Μπαγκλαντές μπορεί λοιπόν έτσι τώρα να εισάγει προϊόντα από το Πακιστάν να τα μεταποιεί και να τα εξάγει με προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν συμφωνία τώρα αν θέλουμε να ενισχύσουμε το Πακιστάν σε βάρος μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Δηλαδή βλάπτουμε και τους εαυτούς μας πλέον και μάλιστα και πριν από την υποβολή του νέου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση των εμπορικών προτιμήσεων. Για μένα το συμπέρασμα είναι συνεχίστε την άμεση ανθρωπιστική ενίσχυση. Γιατί ειδικά στην περίπτωση του Πακιστάν με κάθε μέρα που περνά χάνουμε εμπιστοσύνη σε μας και αξιοπιστία. Δημοκρατίας ο κύριος Μοργκάντη για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η έκθεση αυτή ειλικρινά είναι απαράδεκτη γνωρίζουμε τις τραγικές πλημμύρες που έπληξαν ε, το λαό του Πακιστάν και θεωρώ ότι είναι σωστό να τους βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη τους έχει δώσει ε, μισό δις ευρώ, που δεν είναι και λίγα χρήματα. Αυτές οι εμπορικές προτιμήσεις είναι παράλογες, διότι επικεντρώνονται σε ένα τομέα όπως είναι η κλωσταϊφαντοργία που είναι κυρίαρχο στο Πακιστάν, ενώ στην Ευρώπη σχεδόν καταστράφηκε από τον αγωνισμό των ασιατικών χωρών. Θέλουμε να δώσουμε τη χαριστική βολή στον τομέα της κλωσταεφαντοργίας Εμεί, Εμείς τις Λέγκα του Βορρά δεν το θέλουμε και φυσικά δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Το θέμα αυτό θα πρέπει να περάσει μετά από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο στον ΠΟΕ. Φαίνεται ότι κάποιες χώρες, μεταξύ των ε, οποίων και η Ινδία που αναφέρθηκε, που είναι ιστορικός εχθρός του Πακιστάν, δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν την έγκρισή τους. Θα τη δώσουν μόνο για να έχουν ανάλογες προτιμησιακές ε, ε, συμπεριφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα δεχτούν αυτές τις προτάσεις. Θεωρώ ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπαγορεύεται από το χειρότερο ε, εγωισμό που είναι δυνατόν και ελπίζω να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, το 2010 στο βορειοδυτικό Πακιστάν συνέβησαν από, ε, λόγω των πλημμυρών δηλαδή, τέτοιες καταστροφές που δεν είχαν, δεν προκύψει προηγουμένως από κανέ... οποιαδήποτε άλλη αιτία. Δόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια. Σύντομα η χώρα αυτή θα λάβει το καθεστώς αναπτυσσόμενης χώρας με ειδικό προτιμησιακό καθεστώς σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές. Όμως αυτά δεν έχουν ανακόψει την πρόοδο της, ε, των Ισλαμιστών και μάλιστα σε μια χώρα με πυρηνικό εξοπλισμό. Και οι Αμερικανοί απέτυχαν εκεί παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν διαθέσει. Έτσι λοιπόν η Δύση έχει αποτύχει. Η εκαθάριση του Μπιν Λάντεν έθεσε ωστόσο και ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. Γνώριζε το Πακιστάν την παραμονή εκεί του επικεφαλής της Αλκάιντα. Η γνώση ή η μη γνώση αυτή δεν αλλάζει τίποτε στο ότι με την εκτέλεση του Μπιν ε, Λάδεν παραβιάζεται η κυριαρχία του Πακιστάν. Βεβαίω, τρομοκράτε και άλλοι οφείλουν να άγονται ενώπιον των δικαστηρίων και όχι να εκτελούνται. Περνάμε τώρα στου Ο κύριο ε, Ράγκελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους τον κύριο Μάριο Ντάβιτ του Λαϊκού Κόμματος που δυστυχώς σήμερα δεν είναι παρόν και να πω ότι θεωρούμε ότι η υποστήριξη των θυμάτων των θεομηνιών του Πακιστάν είναι ηθική μας υποχρέωση και γι' αυτό υποστηρίζουμε κάθε μέτρο το οποίο ελήφθη στα πλαίσια δηλαδή της παραδοσιακής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θεωρούμε δε ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για να δοθεί βοήθεια στον κόσμο αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να χρησιμοποιείται ως μέσον για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Διότι αυτό έχει δύο εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις. Αφενός σε βάρος των νότιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος δηλαδή της υφαντουργικής του βιομηχανίας η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης και βεβαίως έχει συνέπειες και στην παγκόσμια οικονομία του ΠΟΕ διότι εάν ανοίξει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο οικονομικό μπλοκ στον κόσμο τις εισαγωγές της για εισαγωγές δηλαδή από το Πακιστάν αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν οφείλουμε να πούμε σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πακιστάν τους τελευταίους 9 μήνες θα πρέπει να καταθέσουμε πιο επικοδομητικές προτάσεις και θα πρέπει να λάβουμε θέση με τροπολογίες να υποστηρίξουμε δηλαδή τις τροπολογίες ώστε εν τέλει να απορριφθεί αυτή η έκθεση και να απορριφθεί η πρόταση κανονισμού μπορούμε να φροντίσουμε να συνεχίσετε να, δίνε, να συνεχίσει να δίνεται η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά όχι με τη μορφή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η έκθεση αυτή για το Κοινοβούλιο ήταν περίπλοκη, καταρχάς γιατί περιλάμβανε αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζονται και το, η έγκριση του ΠΟΕ και η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο είναι διαφορετική από αυτή που απεστέλει στη Γενέβη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν, κατανοούμε ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη κάποιες εμπορικές προτιμήσεις. Ε, αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπόψη και τη ε, συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το τομέα της κλωστοϊφαντεργίας. Ο τομέας στην Ισπανία πλήττεται απευθείας από τις συνέπειες της κρίσης και η έκθεση αυτή μας επέτρεψε να κατανοήσουμε ότι τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίων δεν μπορούν να ε, αντιμετωπιστούν με τον κατεπήγον χαρακτήρα που απαιτούν τέτοιε δράσει. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου για το μέλλον. Ναι, δεχόμαστε τη βοήθεια στο Πακιστάν, αλλά όχι με την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πλήττει τον ε, την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα καθυστερήσει και την εφαρμογή των μέτρων αυτών γιατί εκρεμεί και το κείμενο το οποίο προβλέπεται να εγκρίνει ο ΠΟΕ. Ε, είμαστε λοιπόν εκτός προθεσμιών και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να διατηρήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να την καταψηφίσουμε. Κύριος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Με τη συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού για άλλη μια φορά βρισκόμαστε ενώπιον μια σαφού και επωνίδωση τη διαδικασία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω συνήθω. Διότι μετατοπίζεται σε ανθρωπιστική βοήθεια σε κάτι το οποίο είναι εμπορικά συμφέροντα, είναι επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια υποκριτική διαδικασία που χρησιμοποιεί θεομηνίες που πλήττουν μια χώρα όπως το Πακιστάν για να αποδώσει υποτίθεται δικαιοσύνη ε, στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Σήμερα η δικαιολογία είναι η ανθρωπιστική βοήθεια προς το Πακιστάν. Εχθές ήταν η βοήθεια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο λόγος είναι πάντα ο ίδιος. Να έχουμε εμπορικές προτιμήσεις οι οποίες βοηθούν τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγές. Και όσο και αν ε, προσπαθεί να μας χρυσώσει το χάπι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ρήτρα διασφάλισης που στην ουσία δεν, δεν αλλάζει τίποτα, αυτές οι εμπορικές προτιμήσεις θα καταστρέψουν τον τομέα της κλωσταϊφαντουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από το συγκεκριμένο τομέα ο τομέας ήδη έχει πληχθεί ιδιαίτερα από την αποδυνάμωση του εμπορίου και είναι συγκεντρωμένο σε περιοχές που υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ένδυας και ανεργίας και αυτό σημαίνει ότι γίνονται ακόμα σοβαρότερα τα γεγονότα αυτά όταν βρισκόνται σε μια χώρα όπως είναι η Πορτογαλία που ήδη πλήττεται από μια πολύ σημαντική οικονομική και κοινωνική κρίση που θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από αυτή τη σοβαρή και παράνομη παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην Πορτογαλία το Κοινοβούλιο ενέκρινε είναι ομόφωνα την ε, άρνηση αυτών των εμπορικών προτιμήσεων, διότι πλήττεται ο ευρωπαϊκό κλωστοϊφαντουργικό τομέα και πραγματικά δεν θεωρούμε ότι έχει τίποτα να μα προσφέρει πρώτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μία έκθεση που πίσω από το μανδέα της αλληλεγγύης ουσιαστικά πλήττει τους ίδιους τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι ένα τομέα όπω ο κλωστοϊφαντουργικό, ιδίω για χώρε όπω είναι η Ιταλία, είναι ένα τομέα υψηλή ποιότητα και πρέπει να ανταγωνιστούμε χώρε όπω την Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία και τώρα πλέον και το Πακιστάν που έχουμε εκμετάλλευση των ανθρώπων και πολύ χαμηλού μισθού και δεν λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στι χώρε αυτέ ε, αυξάνεται η παραγωγή και χάνονται θέσει εργασία για την Ευρώπη. Δεν περιμέναμε δεν να μάθουμε τι άποψη έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για το θέμα αυτό. Η Ευρώπη πάντα φαίνεται να δίνει τα μέγιστα για να ε, παραβιάσει τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών της και ελπίζω η έκθεση να καταψεφιστεί. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς και υποστηρίζω την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό του δυνατού. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό της Κομισιόν για την παροχή βοήθειας με τη μορφή των μονομερών εμπορικών παραχωρήσεων υπέρ του πακιστάν. ωστόσο δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις προτάσεις της κομισιόν σύμφωνα με τις οποίες καλούνται να σηκώσουν το βάρος ως επιτοπλίστων δύο βιομηχανικοί τομείς της ένωσης δηλαδή η κλωστοϊφαντουργία και η Βιοϊθανόλη. επισημαίνω ότι η ευρωπαϊκή κλωστοϊφαντουργία δέχτηκε οξύτατες πιέσεις τα τελευταία έτη στην της απελευθέρωση του εμπορίου στο πλαίσιο του παγκοσμίου οργανισμού εμπορίου. κυρίε και κύριοι συνάδελφοι υπήρξα βουλευτή επί τέσσερι ε, θητείε μια περιφέρεια μια περιοχή τη οποία η περιοχή τη νάουσα γνωρίζει σήμερα έναν από του υψηλότερου δείκτε ανεργία σε όλη την ευρώπη και αυτό οφείλεται στι επιπτώσει παγκοσμιοποίηση στην κλωστοϊφαντουργία. όσον αφορά την βιοεθανόλη τονίζω τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ένωση για την ε, νεότευτη αυτή βιομηχανία. δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για δύο βιομηχανικούς κλάδους όπου το πακιστάν εμφανίζεται ιδιαίτερος ανταγωνιστικό. επιπλέον οι εν λόγω παραχωρήσεις δεν συνδέονται με μια ρήτρα αιρεσιμότητας conditionality όπως θα ίσχυε σε περίπτωση που αναγνωριζόταν στο στο πακιστάν καθεστώς gsp σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν. τέλος θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον οι ελόγω παραχωρήσεις θα ωφελήσουν τους ίδιους τους πληρωμα... κατοίκου ε, πλημμυροπαθείς κατοίκους του πακιστάν. επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω και για να μητρηθούν οι αγαθές προθέσεις εδώ μέσα αντιπροτείνω ναι να γίνουν παραχωρήσει αλλά σε άλλα βιομηχανικά προϊόντα γιατί στην, συγκεκριμένα στην κλωστοϊφαντουργία θα ήμασταν εξίσου χρήσιμοι έναντι των πλημμυροπαθών του πακιστάν. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τουλάχιστον να περιοριστούν η χρονική διάρκεια και το εύρος των παραχωρήσεων και να προβλέπονται μέτρα διασφάλισης όπως προτείνεται με τις τροπολογίες του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ο κύριος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι έχουμε την πεποίθηση ότι οφείλουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου του Πακιστάν. Νομίζω όμω ότι το μέσον που προτείνεται κύριε Επίτροπε, είναι λάθο για του εξή λόγου. Πρώτον, δεν αποδεικνύεται ότι οποιασδήποτε εμπορικέ διευκολύνσει θα βοηθήσουν πραγματικά του πλημμυροπαθεί. Αντιθέτω, διαπιστώνεται ότι η κλωστοφαντουργία στο Πακιστάν εδράζεται σε άλλες περιοχές και μάλιστα έχει τα τελευταία χρόνια και σημαντική αύξηση παραγωγής. Άλλη λοιπόν είναι Άλλα, αν λοιπόν θα υποφεληθούν εν τέλει. Δεν βλέπουμε ποιο τρόπο θα ωφεληθούν οι πλημμυροπαθείς. Δεύτερο, δεν μπορώ να κατανοήσω πως μια χώρα η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ε, συνθήκες και τους όρες του GSP+, λαμβάνει τώρα τέτοιες διευκολύνσεις, ενώ άλλες χώρες οι οποίες πληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές, όπως το Μπαγκλαντέ, δεν λαμβάνουν τις προτιμήσεις αυτές. Τρίτο επιχείρημα κύριε Επίτροπε, δεν είναι προσέγγιση αλληλεγγύης, διότι η επιβάρυνση που θα βαρύνει την Ευρώπη είναι μονομερής σε ορισμένους τομείς και ορισμένες χώρες. Εάν θέλουμε και πρέπει να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε αλληλεγγύως με συμμετοχή όλων των χωρών και όλων των ενδιαφερομένων. Να δώσουμε εν τέλει δηλαδή άμεση βοήθεια στα θύματα των πλημμυρών. Αυτό θα ήταν το σωστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν αρκεί να εκφράζουμε την λύπη μας για τις θεομηνίες Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Ένωση δεν περιορίστηκε σε αυτό, αλλά αμέσω χορήγησε βοήθεια. Το μέλλον του Πακιστάν είναι σημαντικό για ολόκληρο τον κόσμο και για την Ευρώπη. Είναι σημαντική χώρα, ιδιαίτερα ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και έρχονται αρκετοί μετανάστες στην Ένωση από εκεί. Μέχρι τώρα όμως η Ένωση δεν έχει εκφράσει καμία συγκεκριμένη πολιτική για το Πακιστάν. Αυτό το σύστημα εμπορικών προτιμήσεων δεν βασιζόταν σε συγκεκριμένα στοιχεία, δεν μπόρεσε η Κομισιόν καν να μας το δικαιολογήσει. Κατά τη συνάντησή του με τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Τα οι δεν είναι σίγουρο ότι θα ωφεληθούν από αυτό μόνο δύο συμφέροντα έχει η Ένωση στη σχέση της με το Πακιστάν, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και από την άλλη την ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό πρέπει να βασίζεται όπως και παντού στον νόμο. Αν λοιπόν δεν έχουν σταθεί στόχο οι προτάσεις αυτές, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Πρέπει να υπάρξει ολόκληρο πρόγραμμα υποβοήθησης της ανάπτυξης της χώρας με τον όρο όμως αν θέλει στενότερες σχέσεις το Πακιστάν με την Ένωση να μπορεί να αποδείξει ότι πραγματικά ε, είναι κράτος δικαίου και καταπολεμεί την τρομοκρατία. Συνολικά όμως, όχι προτάσεις που να περιορίζονται σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουσα πρόταση πρέπει να απορριφθεί και η κυρία Άστον να υποβάλει νέα συνολική πρόταση με όρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι 8 μήνες τώρα από τότε που το Συμβούλιο πρώτο πρότεινε μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυροπαθών και δυστυχώς ακόμη τα συζητάμε και δεν τα εφαρμόζουμε. Γιατί χρειαζόταν οι προτάσεις αυτές. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ βοήθειας και εμπορικών σχέσεων. Είναι σημαντική και η βοήθεια για το Πακιστάν, αλλά αυτή η εμπορική δέσμη στόχευε να δώσει κίνητρα στους επιχειρηματίες για να συνεχίσουν ή να αρχίσουν την ανάπτυξη της χώρας γιατί αντιμετώπισαν και αυτοί οι προβλήματα με τις πλημμύρες. Βέβαια ο κύριος τομέας που επλήγει αφορούσε όντως την υφαντουργία αλλά δεν ήταν ο μόνος. τα κίνητρα για την ανοικοδόμηση της υφαντουργίας θα έπρεπε να βασίζονται στις αγορές από την Ένωση, να δουν οι επιχειρηματίες δηλαδή ότι υπάρχει αγορά για τα προϊόντα τους. Η ιδέα ρήτρα ασφαλείας που ισχύει μόνο για ένα χρόνο είναι κάτι χωρίς κανένα νόημα. Επίσης λυπάμαι γιατί η Ινδία δεν υποστήριξε στον ΠΟΕ ανάλογα μέτρα για το Πακιστάν. Ελπίζω η λεγόμενη δημοκρατία του κρίκετ να αποφέρει τελικά ε, διπλωματία του κρίκετ, να αποφέρει τελικά κάποια αποτελέσματα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον. Ευχαριστώ. πρώτη κυρία Ζαμπόρσικα για ένα λεπτό. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Βλέπω ότι το θέμα αυτό διαιρεί τους βουλευτές μας. Παρόλα αυτά και παρόλα όσα άκουσα, συμφωνώ με το Συμβούλιο. Είμαι μέλος της Επιτροπής Αναπτύξεως και νομίζω ότι η πτυχή αυτή της άμεσης δηλαδή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τέτοιες ε, περιπτώσεις θεομηνιών είναι απαραίτητη. Ωστόσο δεν είναι επαρκής. Καλύτερα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Γι' αυτό και θεωρώ σωστή την άρση των ε, δασμολογικών φαγμών για τις εξαγωγές του Πακιστάν και για μια περίοδο που να επιτρέψει το Πακιστάν να ξεπεράσει τα προβλήματα. Η προσέγγιση αυτή είναι χρήσιμη. Και αν αυτό αποδειχθεί, ίσως πρέπει να επανεξετάσουμε και να επανακαθορίσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί ο μεγάλος ανταγωνισμός είναι η Κίνα στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και άλλοι προηγουμένως, βλέπουμε ότι οι εμπορικές αυτές προτιμήσεις που χορηγούνται στο Πακιστάν δεν θα αποτελέσουν λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πλημμυροπαθών. Το εμπόριο δεν είναι το καταλληλότερο μέσο για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Συμφωνώ βέβαια ότι μπορεί αυτά τα μέτρα συγκεκριμένα να μην αφορούν όλους τους πλημμυροπαθείς Ορισμένους όμως τουλάχιστον τους αφορούν η διεθνής βοήθεια και το εμπόριο πρέπει να συνδυαστούν. Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Όταν χορηγούμε βοήθεια ή προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις με ορισμένες χώρες δεν το κάνουμε μόνο για το συμφέρον μας αλλά και για να τις εξυπηρετήσουμε. Οι πλημμύρε το τελευταίο καλοκαίρι στο Πακιστάν ήταν πραγματικά σοκ και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα για να συνδράμει τους ε, ε, εκατομμύρια Πακιστανών και φυσικά η βοήθεια θα πρέπει να γίνεται χωρίς ε, πολιτικές συνέπειες. Τα μέτρα αυτά που προτείνουμε αυτή τη στιγμή είναι διαφιλονικούμενα και για την περιοχή αλλά και για το Πακιστάν. Η σύλληψη, ο θάνατος του Οσάμα Μπιν Λάνταν και το γεγονός ότι βρισκόταν στο Πακιστάν δείχνει ότι το Πακιστάν ε, είναι αμφιβολιγόμενη χώρα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ουσιαστικά θα ανταμείψουμε την κυβέρνηση του Πακιστάν γιατί δεν έδρασε στον τομέα αυτό. Επίσης, το Μπαγκλαντές, μια χώρα που πλήχθηκε και αυτή από πλημμύρε θα πληχθεί και από το ανταγωνισμό, ιδίω στον τομέα τη κλωσταβεφαντουργία. Αυτό που δέχομαι είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεπτικά το θέμα αυτό, ε, ιδίω για όλου του λόγου που ανέφερα στην ομιλία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η υποβληθήσα πρόταση αποτελεί επίθεση κατά της ευρωπαϊκής κλωστήφαντουργίας. Ωστόσο, να πω και άλλο επιχείρημα. Απελευθέρωση από ε, δασμούς πρέπει να συνδέεται οπωσδήποτε με τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θυμίζω εκεί την μοίρα των χριστιανών, θυμίζω επίσης τι μοίρα επιφυλάσσεται σε όσους θεωρηθεί ότι βλασφημούν το Ισλάμ. Αυτά τα διαπιστώνει κανείς καθημερινά. Το επιχείρημα λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό, με τις προτιμήσεις αυτές θα καταπολεμήσετε τους ριζοσπάστες εκεί, δεν το πιστεύετε τους ίδιους ο ίδιος. Για βασικά θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πράττει τίποτε. Δεν, είχατε, δεν σας έχουμε σημειώσει για το Catch the Eye αλλά αν μου υποσχεθείτε, αν μου δώσετε το λόγο σας ότι θα τη σηκώσει το χέρι σας, θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά κροκοδίλια, είδαμε μάλλον πολλά κροκοδίλια δάκρυα σήμερα από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις 180 μοίρες αντίθετες από αυτές που ε, εκφράζουν συνήθως. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και παλαιότερα. Μας διαβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει κάνει προσεκτική επιλογή των προϊόντων ώστε να μην συγκρούονται με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Μήπως άραξε τίποτε εδώ. Μας ρώτησαν γιατί τα εφάσματα από το Πακιστάν. Μα διότι για αυτούς είναι σημαντικό εξαγώγημο προϊόν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βρουν κάτι άλλο μέσα σε λίγους μήνες. Είχαμε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το εάν θα ωφεληθούν τελικά οι πλημμυροπαθείς. Το συζητήσαμε αυτό όταν πήγαμε στο Πακιστάν και ακούσαμε ευθέως από Πακιστανούς βουλευτές ότι θα ωφελήσει την βιομηχανία στις ίδιες τις εκλογικές τους περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το μήνυμα που θα δώσουμε εάν δεν υποστηρίξουμε τα μέτρα αυτά. Ο ο uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήμουν παρόν στην έναρξη της συζήτηση. Μόλις έφτασα από τις Βρυξέλλες αεροπορικός και ήσασταν και λίγο νωρίτερα με το πρόγραμμα και αυτό φυσικά είχε ως συνέπεια να καθυστερήσω εγώ. Interventions that been... Σημείωσα όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία. Καταρχάς, δεν συζητάμε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Έχω την εντύπωση ότι πολλές από τις παρεμβάσεις ε, ξεκίνησαν από αυτή την προϋπόθεση, ότι αυτή είναι μια μορφή ε, συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της ερεσιμότητας, ε, της βιωσιμότητας ε, και δεν θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη εδώ, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο σαφέστατα είναι χρονικός περιορισμένο. Δεύτερον, δεν συζητάμε σύστημα γενετευμένων προτιμήσεων. Ε, αυτό θα το κάνουμε στο μέλλον και στη διάρκεια της συζήτησης θα δούμε ποιες χώρες μπορούμε να συμπεριλάβουμε και ποιες όχι. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσε τις πλημμύρες στο Πακιστάν. Είναι χρονικώς περιορισμένη για δύο χρόνια με δυνατότητα να παραταθεί για ένα ακόμα έτος. Η δυνατότητα παράτασης ε, Συγγνώμη, το γεγονό ότι ε, προτάθηκε να είναι μόνο για ένα χρόνο, κατά την άποψή μου δεν είναι λογικό. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και γιατί τώρα χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από τις πλημμύρες. Ακριβώς επειδή Εισήχθη το αίτημα απαλλαγή ε, στον ΠΟΕ, αλλά στον ΠΟΕ υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τις γείτονες χώρες του Πακιστάν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας τις κατονομάσω και προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Νομίζω ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και στις επόμενες εβδομάδες ε, θα δούμε τι συνέπειες ε, υπάρχουν σε σχέση και με τα πρόσφατα γεγονότα στο Πακιστάν. Ε, επαφίεται στον ΠΟΕ το κατά πόσον θα δώσει απαλλαγή και φυσικά η δυνατότητα απαλλαγή πρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα. Δεν, ομόφωνα. Δεν μπορούμε να πιέσουμε το θέμα αυτό στον ΠΟΕ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα προκειμένου να περάσει το θέμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και εδώ δεν μιλάω ως ε, όπως ακούσαμε ε, από κάποιον από τις προελίσσαντες για κροκοδίλια δάκρυα και για φρούδες υποσχέσεις. Ε, αυτά που ακούσαμε όμως σήμερα δεν συνάδουν απαραίτητο με αυτά που ακούσαμε στο παρελθόν. Και αυτό δεν έγινε διότι έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και γιατί δεν υπάρχει ακόμα η απαλλαγή από τους δασμούς. Ε, δεν έχει αλλάξει γι' αυτό το λόγο το επιχείρημα. Εξ αρχής υπήρχε η συζήτηση για το κατά πόσον είναι υπέρ των ανθρώπων που πλήχθηκαν από τις πλημμύρες ε, το μέτρο αυτό. Μερικώς είναι. Εξ αρχής ε, υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαμε ανθρωπιστική βοήθεια ε, της τάξης των 480 εκατομμυρίων ευρώ. Τα επιχειρήματα είναι τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ξαφνικά θα πρέπει να αλλάξουμε προς άλλη κατεύθυνση άλλη γραμμή πλεύση. Ε, γνωρίζουμε τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν με τον τομέα της κλωστοϊφαντουργία στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ρήτρα διασφάλισης, προτείνεται μια τέτοια ρήτρα και νομίζω ότι επαρκεί προκειμένου να αντισταθμίσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε γενικέ γραμμέ, νομίζω ότι το θέμα είναι σαφέ ε, και θα πρέπει να δείτε αν είστε υπέρ ή κατά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε υπέρ και για, από το οπτικό πρίσμα τη οικονομική ανάπτυξη του Πακιστάν και από το οπτικό πρίσμα των θεμάτων ασφαλεία που έχουν προκύψει για το Πακιστάν. Θεωρώ ότι θα ήταν μοιραίο σφάλμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην αδράξει τη δυνατότητα και να υπερψηφίσει το θέμα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. ο κύριο Μορέιρα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε de Gucht. Βεβαίω ήρθατε ε, με κάποια καθυστέρηση, αλλά εγκαίρω για να μπορέσετε να ε, πείτε την τελική σα άποψη. Θα ήθελα τώρα να κάνω δύο παρατηρήσει. Αφενό, η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχει μια διαίρεση στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, όπως επίσης και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις ίσως ορισμένες να μην είναι σκόπιμες θα δούμε αύριο τι άποψη θα εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, καταλήγοντας, επιτρέψτε μου δύο ακόμη σχόλια. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ότι προσπάθησε να μπλοκάρει την εξέλιξη της ε, υπόθεσης αυτής. Βεβαίως, εκκρεμεί ακόμα η απαλλαγή από πλευράς ΠΟΕ. Δεν μπορεί να προχωρήσει λοιπόν η δική μας προσπάθεια. Παρ' αυτά εμείς εργαστήκαμε και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε και λάβαμε υπόψη και όλες τις τροπολογίες και τις τροπολογίες που υπεβαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει βεβαίω το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλία, κατέθεσε την πρόταση και μετά καταθέσαμε πρόταση σχετικά με την απαλλαγή από, το ΠΟΕ, αλλά, από αλλά δεν συμπίπτουν οι προτάσεις Τη Επιτροπής με το Κοινοβουλίο. Έχουμε και το συμβασμό του Συμβουλίου που επίσης αποκρίνει από την πρόταση τη Επιτροπή Πάντω, αυτά δεν τα θεώρησε η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου ως εμπόδιο. Προχώρησε, επεξεργάστηκε το κείμενο και ψηφίστηκαν, ψηφίστηκαν όλες οι τροπολογίε και του Συμβουλίου και της Κομισιόν. το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο σημερινής διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδία.